Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στην απογευματινή μας συνεδρίαση. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς ε, και είναι τιμή μας που είναι εδώ ο υπουργό ε, της ε, Σουηδίας, χώρας που ασκεί την εκπεριτροπής Προεδρία του Συμβουλίου. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η βιογραφία σας. Τη διάβασα προσεκτικά. Είστε οδοντίατρος. επιστήμων θα μου πείτε. Ναι. Και ενδιαφέρεστε, σας αρέσει το σκι, όπως και εμένα. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι είστε υπουργός εμπορίου κατά μια στιγμή όπου ο κόσμος προσδοκά σε μια συμφωνία στα πλαίσια του γύρου της Ντόχα και στον ΠΟΕ, τη στιγμή που ο κόσμος αντιμετωπίζει αυτή την οξία οικονομική κρίση, οι δυνατότητες που προσφέρει το εμπόριο για την διέξοδο από την κρίση είναι πολύ σημαντικές, οπότε τα θέματα αρμοδιοτήτως μας, το εμπόριο δηλαδή, δοσμολογικά εμπόδια και ε, όλα τα σχετικά είναι πολύ σημαντικά. Θα καθορίσουν πολλές μελλοντικέ εξέλιξεις. Καλώς ήρθατε και ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που έχετε να μας πείτε. Thank Ευχαριστώ, Ρόμπετ. Κυρίε και κύριοι, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι μεγάλη τιμή μου που βρίσκομαι εδώ για να παρουσιάσω την εμπορική πολιτική της Προεδρίας και τις προτεραιότητες της για το δεύτερο ημίση του 2009. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα την ε, Επιτροπή σας για τον ρόλο που διαδραματίζεται στον καθορισμό της κοινή μα κοινής μας εμπορικής ε, πολιτικής. Σας ενθαρρύνουμε να συνεχίσετε το έργο σας και κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας. Ομοίως θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Τσεχική και Γαλλική Προεδρία για το θαυμάσιο έργο τους και την αγαστή συνεργασία που είχαμε. Η εμπορική πολιτική είναι δυνατότητες και προκλήσεις, είναι παράγοντας ε, σφυριλάτησης ε, ε, καλύτερων συνθήκων για τους Ευρωπαίους πολίτες και ένα κοινά αποδεκτό παγκόσμιο εμπορικό σύστημα είναι επωφελέ για όλου. Επίση, η εμπορική πολιτική μπορεί να συνεισφέρει στου στόχου τη Ένωση για την αηφόρο ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου δηλαδή και του θέματων, θεμάτων του, όπως το κλίμα και το περιβάλλον. Καλούμεθα λοιπόν να αντιμετωπίσουμε επιτυχώ αυτέ τι προκλήσει για το όφελο των πολιτών που έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν την ε, πραγματικότητα της ευρωπαϊκής ε, Δύο λόγια για την κρίση και το παγκόσμιο εμπόριο. Αντιμετωπίζουμε μία από τις σοβαρότερες οικονομικές και δημοσιονομικές κρίσεις των ε, σύγχρονων καιρών. Το παγκόσμιο ΑΕΠ θα είναι αρνητικό ε, για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μείον 5% συνολικά σύμφωνα με την Παγκοσμία Τράπεζα. Παρόλο που έχουμε δει κάποιες αχτίδες φωτός στην άκρη του τούνελ, παρόλο που κάποιες οικονομίες από ό,τι φαίνεται βγαίνουν από την ε, κρίση δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε βεβαίως διότι η πρόοδος αυτή είναι έθραστη και οι προκλήσεις είναι υψηλότατη ανεργία και πολύ σημαντικά δημοσιονομικά ελλείμματα. Επίσης η ανάκαμψη στην Ευρώπη από ό,τι φαίνεται θα καθυστερήσει σε σχέση ε, με τις... Ε, ε, η ανάκαμψη θα καθυστερήσει σε σχέση με τις ΗΠΑ και άλλες περιοχές του κόσμου. Και αυτό θα έχει βεβαίως αρνητικές συνέπειες. Το παγκόσμιο εμπόριο επλήγει λοιπόν σκληρά από την παγκόσμια κρίση. Γενικά το εμπόριο προβλέπεται ότι θα συρρυκνωθεί κατά 10% το 2009. Η φυστάμενη επιβράδυνση έχει πλήξει όλες τις χώρες, παρόλο που οι αναπτυσσόμενες πλήντονται περισσότερο με μείωση των εμπορικών τους ρόλων κατά 14%. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σημειώνει ότι παρά τις, ε, ε, ε, τις δειλές προβλέψεις για πρόοδο, η προοπτική για την εξωτερική ζήτηση για την περιοχή του ευρώ θα συνεχίσει να συρρυκνούνται. Ως συνέπεια των κρίσεων αυτών οι προστατευτικέ τάσεις έχουν αναφηθεί εκ νέου και αυτό είναι ενισχυτικό ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εθνικιστικές διατάξεις, τι δημόσιες ε, προμήθειες, νέες κρατικές επιδοτήσεις, νέες δασμολογικά ε, και άλλα ε, εμπόρια, εμπόδια στο εμπόριο. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη πίεση επιστροφή στον προστατευτισμό. Αυτό θα ενταθεί ως φαινόμενο όσο ανεβαίνουν τα επίπεδα, τα ποσοστά της ανεργίας. Νέα μέτρα διακριτικής μεταχείρισης τρέβλωσης του ανταγωνισμού θα πλήξουν την προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας και είναι σημαντικό να έχουμε κατά ότι το εμπόριο δεν φταίει, δεν είναι υπεύθυνο για την κρίση. Οι ανοιχτέ αγορές και ένα δυνατό, ισχυρό, πολυμερές εμπορικό σύστημα είναι προϋποθέσεις για την οικονομική ανάκαμψη μαζί όλοι εσείς ως μέλη αυτής της Επιτροπής, εμείς ως Προεδρία έχουμε σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε. Να διστοποιήσουμε τους πολίτες για τη σημασία αυτής της πολιτικής που θα πρέπει να την υποστηρίξουν. Αλλά αυτό θα γίνει μόνο αν, καταφέρουμε να εξηγήσουμε τα ωφέλη της εμπορικής, της εμπορικής αυτής της πολιτικής, ιδιαίτερα σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς. Η πρωτοβουλία του Πασκάλ Λαμή είναι πολύ σωστή διότι ε, η διαφάνεια και η πίεση που ασκείται στους ε, ισότιμους ε, εταίρους μας είναι κάτι πολύ σημαντικό και το Δελτανιτάφ και ο ΣΑΚ και η Κεντρική Τράπεζα έχουν, και η Παγκόσμια Τράπεζα συγγνώμη, έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην, στο ίδιο πλαίσιο. Στενή συνεργασία λοιπόν και συντονισμό μεταξύ των διεθνών αυτών βημάτων είναι ζωτική σημασία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει ε, την παρακολούθηση των πραγμάτων από την πλευρά της, το monitoring της δηλαδή, επί τη βάση των στοιχείων ε, που θα συλλέγει ε, από τα επιτελεία της που προέκυψαν από την εταιρική σχέση μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ανοίξουν οι αγορές και να έρθουν τα δεσμολογικά εμπορία στις τρίτες χώρες. Η εταιρική σχέση είναι ένα κοινό πρόγραμμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών και της επιχειρηματικής κοινότητας που γίνεται και στις Βρυξέλλες αλλά και επιτόπου σε τρίτες χώρες η συνδυασμένη ισχύ 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της, επιστημον... κοινότητα επιχειρηματικής κοινότητας μας δίδει περισσότερα όπλα να άρουμε τα δασμολογικά εμπόδια σε άλλες χώρες. Κατά τη διάρκεια των τσεχικών, γαλλικών και τώρα τη Σουηδικής προεδρία, έχει τεθεί περισσότερη ε, έμφαση στον καθορισμό προτεραιοτήτων, στην άρση των δασμολογικών εμπορίων και στον καθορισμό στρατηγική για την καταπολέμηση αρνητικών φαινομένων σε σημαντικές χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Ιαπωνία, η Βραζιλία. Δεδομένου αυτών των συνδικών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει τον ηγετικό του ρόλο, να συνεχίσει να έχει τι αγορέ ανοιχτέ και να αποφεύγει πάση θυσία προστατευτικέ δράσει. Ο οικονομικό εθνικισμό βεβαίω θα πρέπει να αποφευθεί. Ε, ακόμα και όταν παίρνει μορφή διαφορών πακέτων ε, ανάκαμψη, ε, υποστήριξη. Θα πρέπει λοιπόν παγκόσμια αυτό να είναι η ε, αρχή που θα ακολουθούμε. Η ενότητα και η συντονισμένη δράση εντός της ενώσεως είναι ε, το καλύτερο εργαλείο, το καλύτερο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές αυτές προκλήσεις και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βγει από την κρίση δυναμωμένη. Περνάω τώρα στην Τόχα. Η ολοκλήρωση του γύρου της Ντόχα είναι η πρώτη, δεύτερη και τρίτη προτεραιότητά μας. Όλα τα μέλη του ΠΟΕ και ιδιαίτερα οι αναπτυσσόμενες χώρες θα δρέψουν πολύ σημαντικούς καρπούς σε αφορά την πρόσβαση στις αγορές και άλλα θέματα. Επίσης, η αξία θα έλεγα του γύρω της Δόχα έχει αυξηθεί ε, πολύ περισσότερο λόγω ε, του ασφαλιστικού ε, του δικτύου ασφαλείας που θα αποτελέσει έναντι προστατευτικών μέτρων. Ευτυχής ολοκλήρωση του γύρου της Ντόχα μέχρι το 2010 θα δώσει ένα οικονομικό κίνητρο και θα προωθήσει ε, τα μέτρα ένταξης των αναφιόμενων οικονομιών στο πολυμερές ε, παγκόσμιο σύστημα. Αποτυχία του γύρου της Ντόχα θα είναι μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Έτσι πιστεύω ότι ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΕ, ο κύριος Πασκάλ Λαμή, ε, θα είναι σε θέση σύντομα να καλέσει μια συνάντηση πολιτικό επίπεδο στη Γενέβη για να ε, ε, συμφωνηθούν εφαρμοστικές λεπτομέρειες για την πρόσβαση στην αγορά για τα αγροτικά προϊόντα αλλά και τα υπόλοιπα. Θα πρέπει να έχουμε μια σαφή βεβαίως ιδέα για τις συνιστώσεις ε, που θα συναποτελούν το τελικό πακέτο. Και βεβαίω να συνδευτεί όλη η διαδικασία με μια καταληκτική προθεσμία. Θα πρέπει να συνεχιστούν δε οι συζητήσει σε ένα ευρύ φάσμα πολύ σημαντικών θεμάτων που θα αποτελέσουν κομμάτι ε, του λεγόμενου single undertaking, της τελικής δηλαδή συμφωνίας ε, και της αρχής ότι τίποτα δεν συμφωνείται μέχρι να συμφωνηθούν τα πάντα η σύμπλευση των Αμερικανών είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις πιέσεις ε, επί της νέας Αμερικανικής κυβέρνησης ε, να ανοίξει τις αγορές της, βάλει ελεύθερο εμπόριο και να ολοκληρώσει ε, τις βασικές προτεραιότητες στα πλαίσια του γύρω της Ντόχα. Στο Πίτσπερκ, στην συνάντηση της ομάδος των 20, ελπίζω να δοθεί μια νέα όθηση στην προσπάθεια αυτή που θα συνεχιστεί το φθινόπωρο. Οι πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες είναι βεβαίως ο προτιμητέος τρόπος, ε, η προτιμητέα άγουσα. Όμως και οι διμερείς εμπορικές συμφωνίες είναι παραπληρωματικές ε, των πολυμερών και μπορούν πολλές φορές να προωθήσουν αποτελεσματικά τα συμφέροντα της Ένωσης στις ε, αγορές. Και υποστηρίζω τα λεγόμενα της Επιτρόπου Άστον υπό την έννοια αυτή. Περιφερειακές και διμερείς όμως συμφωνίες ποτέ δεν μπορούν να υποκαταστήσουν πολυμερείς συμφωνίες. Προετοιμάζουν απλώς το δρόμο, αποτελούν το πρώτο βήμα στο δρόμο που οδηγεί σε μια πολυμερή συμφωνία. Σημαίνει ότι οι χώρες αυτές ε, και αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες ε, επιδιώκουν κοινούς στόχους που όμως δεν είναι πάντα δυνατόν να εφαρμοστούν ε, από όλους την ίδια στιγμή. Η μεγαλύτερη πρόσβαση στις αγοράς, αναφιόμενες οικονομίες, Ασία, Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή, είναι πολύ σημαντική και την ανταγωνιστικότητα της ίδιας της Ένωσης. Μέσω της ε, βελτίωσης ε, του κλίματος στο οποίο κινούνται οι επιχειρήσεις και γίνονται οι συμφωνίες αυτές μπορούμε να βοηθήσουμε στη μείωση της υποανάπτυξης και της φτώχειας στις ε, αναπτυσσόμενες ε, χώρες. Έτσι, η οικονομική συνεργασία μπορεί να υποστηρίξει ευρύτερη πολιτική συνεργασία και να ε, αντιμετωπίσει και θέματα που αφορούν την παγκόσμια ασφάλεια. Ας πω δύο λόγια τώρα για το που βρισκόμαστε προς το παρόν για ορισμένες από τις ε, διαπραγματεύσεις FTA της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας ξεκινήσω με τη, με Νότια Κορέα. Ε, μια συμφωνία με την ε, Νότια Κορέα τον πέμπτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ένωσης αποτελεί προτεραιότητα. Το, η συμφωνία αυτή έχει ενδυνάμει να προσφέρει πολλά ωφέλη και στους εισαγωγείς και στους εξαγωγείς μέσω της άρσης ε, των ε, δασμών, των εμποδίων στην παροχή υπηρεσιών και την πώληση ε, αγαθών. Χαιρετίζω το γεγονός ότι τώρα έχουμε επιτάπητο ένα τελικό συμβαστικό πακέτο και ελπίζω ότι η συμφωνία θα συναυθεί και επίσημα όσον ούπο, ούτω ώστε να καταδείξουμε ότι είμαστε σοβαροί σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει του ελεύθερου εμπορίου και ότι θέλουμε να έχουμε τέτοιου επαφέ. Ινδία δεν διαφαίνεται συμφωνία. Όμως ε, με τη νέα Ινδική κυβέρνηση νομίζω ότι θα έχουμε μια νέα όθηση στη συζήτηση ε, κατά τη διάρκεια του 2010 σε σχέση με τις χώρες ΑΣΕΑΝ. Μέσω και βράχη πρόθεσμα θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη δυνατότητα ε, προώθησης ε, των συζητήσεων με τις διάφορες χώρες ΑΣΕΑΝ ανάλογα με την ε, περίπτωση, ανάλογα με τη δυνατότητά τους δηλαδή να συνάψουν αυτές τις συμφωνίες με την Ένωση, έχοντας βεβαίως κατά νου και το συνολικότερο στόχο που αφορεί όλη την περιοχή ως δέσμη, ως μία περιφέρεια. Επίσης και με τις χώρες του Συμφώνου των Άνδεων επιδιώκουμε ε, επίλυση των προβλημάτων, όπως αυτό της μπανάνας, που βεβαίως δεν εξαρτάται μόνο από εμά, αλλά και από τις ιστορικές διαφουλεύσεις ε, των ε, χωρών που δεν συμμετέχουν όλες αυτές, όπως η Βολεβία και το Εκουαδόρ. Γι' αυτό εμείς θέλουμε να ασκήσουμε πάσα πίεση προς την κατεύθυνση αυτή οι συμφωνίε σύνδεση με την Κεντρική Αμερική. Έχουν ξεκινήσει και καλά κρατούν. Όμω οι ατυχεί εξελίξει ε, στην Ονδούρα ε, μα αναγκάσαν να αναβάλουμε τι σχετικέ ε, συζητήσει. Θα πρέπει λοιπόν να επιληθεί το πρόβλημα πριν μπορέσουμε να επανακάμψουμε στις συζητήσεις. Διαπραγματεύσεις FTA με το GCC έχουν ανασταλεί από τον περασμένο Δεκέμβριο λόγω δύο ανοιχτών θεμάτων. Το ένα αφορά πολιτικές ρήτρε και το άλλο το θέμα των εξαγωγικών δασμών. Εμείς ως Προεδρία θα καταβάλουμε πάσα προσπάθεια για να διευκολύνουμε την πρόοδο και την ευτυχή ολοκλήρωση αυτών των διαπραγματεύσεων. Παρ' όλα αυτά, για να το επιτύχουμε αυτό, και τα δύο μέρη θα πρέπει να επιδείξουν ελαστικότητα και συμβαστικό πνεύμα. Ε, συμφωνίες ΕΠΑ οικονομικές εταιρικές, ε, συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Είναι πολύ σημαντικές για τις χώρες ε, ε, του Ειρηνικού και της Καραϊβικής, τις χώρες ΑΚΕ. Μακρές μεταβατικές περίοδοι και ε, ανάληψη δεσμεύσεων από τις χώρες αυτές ε, συνοδεύονται από συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν την εφαρμογή των συμφωνιών αυτών. Ο βραχυπρόθεσμος, αυτός είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος. Ο βραχυπρόθεσμος στόχος είναι η υπογραφή και επικύρωση ε, των ενδιάμεσων ΕΠΑ. Παρ' όλα αυτά ο βασικός στόχος θα πρέπει να μείνει αναλύωτος. Πρέπει δηλαδή να έχουμε συμφωνίες περιφερειακής συνεργασίας συνολικές και σφαιρικές γιατί μόνο αυτές μπορούν να ε, αξιοποιήσουν το δυναμικό που υπάρχει για, τις, ε, για τη βελτίωση των εμπορικών ιερών ροών από και προς τις χώρες αυτές, ιδιαίτερα τώρα σε αυτούς τους καιρούς οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει ε, βαρέως τις χώρες αυτές και ιδιαίτερα το εμπόριό τους. Με χαρά σημειώνω ότι υπάρχει σημαντική βελτίωση του κλίματος εντός των Εντο του οποίου γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Έτσι έχουμε ήδη δει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα αυτού του νέου θετικού κλίματος. Χαιρετίζω ιδιαίτερα το γεγονός ότι η ανατολική εταιρική σχέση ε, της Ένωσης ξεκίνησε στην Πράγα στις 17 Μαΐου. Έχουμε πλέον ε, τη δυνατότητα διμερών ε, συμφωνιών μεταξύ Ένωσης και κάθε μίας από τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Ουκρανία, Μολδαβία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, και ε, ο στόχος είναι να έχουμε ουσιαστικές ε, FTAs όταν οι χώρες αυτές είναι έτοιμες. Περισσότερη ανάπτυξη της εταιρικής μας εταιρικής σχέσης είναι προτεραιότητα για την ε, Προεδρία μας. Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος που βρίσκεται στην άμεση γειτονιά μας. Έχει γίνει πρόοδος στα πλαίσια των FTA, αλλά όχι τόσο όσο θα επιθυμούσαμε διότι υπάρχει και μεγαλύτερη οικονομική πίεση τώρα πλέον με την κρίση. Επίσης υπάρχει μια σειρά διμερών προβλημάτων που αφορούν δασμολογικά μέτρα που έχουν λάβει οι Ουκρανοί και που έχουν επιβαρύνει το κλίμα. Ρωσία. Η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη οικονομία εκτός ΠΟΕ. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος ε, εταίρος της Ρωσίας. Η προσχώρηση της ε, Ρωσίας στον ΠΟΕΛ ως εκ τούτου θα είναι προς ε, ε, όφελος όλων. Όσο περισσότερα, όσο πιο γρήγορα γίνει η προσχώρηση αυτή, τόσο πιο γρήγορα θα δρέψουμε τους καρπούς αυτής της προσπαθίας. Οιαδήποτε καθυστέρηση θα ήταν λυπηρή. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά πρέπει να είμαστε να σταθούμε ισχυροί και να μην κάνουμε παραχωρήσεις επί των αρχών που έχουμε θέσει. Θέλουμε λοιπόν η Ρωσία να κινηθεί προς ολοκλήρωση της ε, υποψηφιότητάς της ε, σε ένα όχι απότερο μέλλον. Η προσχώρηση στον ΠΟΕ της Ρωσίας θα αποτελέσει προϋπόθεση και θα προετοιμάσει τον δρόμο για ομαλότερες διπλωματεύσεις... για εμπορικά θέματα και θέματα που αφορούν τις επενδύσεις ε, στην Ρωσία γιατί έτσι μόνο θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την βαθιά αλλά και πολύπλοκη σχέση που έχουμε με την Ρωσία. Η ημερομηνία στόχος 2010 για την ε, δημιουργία ενός χώρου ελευθερού εμπορίου ευρώ, στην ε, ευρωμεσογειακή περιοχή. Έχει ήδη συμφωνηθεί. Αυτό που μένει είναι να συμφωνήσουμε ε, εφενός φιλουπορίας. πορείας και αυτό ελπίζω ότι θα γίνει στην ε, Υπουργική Διάσκεψη κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας κατά πιθανότητα τον Οκτώβριο. Οι διατλαντικές εμπορικές σχέσεις είναι, ε, αφορούν ε, το μεγαλύτερο μακράν όγκο εμπορικών ροών και μία πρόοδος στον τομέα αυτό θα είναι υποφελής και για την Ένωση και για τη ΣΥΠΑ παρά κάποια πρόοδο. Έχει αποδειχτεί ότι είναι δύσκολο το θέμα και χρειάζεται αναζωπήρωση και αναζωογόνηση των προσπαθειών μας. Προς αυτό το σκοπό, το Οικονομικό Διατλαντικό Συμβούλιο που θα συναντηθεί τον Οκτώβριο είναι κεφαλαίο σημασίας. σημασία. Ως πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ε, προσπάθεια αναφύσης νέων δασμολογικών και εμπορικών εμποδίων και όχι στην επίλυση των υπαρχόντων, γιατί αυτό θα αποδειχθεί, αν όχι ανεπίλητο, εξαιρετικά δυσεπίλητο πρόβλημα. Να προλάβουμε λοιπόν την αναφύγηση νέων εμποδίων. Ο μακροπρόθεσμος στόχος θα πρέπει να είναι μια, ε, ευρω... μια διατλαντική αγορά απαλλαγμένη από εμπόδια. Και εδώ χαιρετίζω ιδιαίτερα το γεγονό ότι θα ξεκινήσουν οι και με τον Καναδά για μια συνολική συμφωνία εμπορική και οικονομική φύσεω. Και αυτό κατά τη διάρκεια τη ε, Σουηδική Προεδρία. Κίνα. Η Κίνα είναι η λιδία λίθο ε, της προσπάθειας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εμπορικής πολιτικής. η επερχόμενη διάσκεψη κορυφής ε, αλλά και η μεταγενέστερη το φθινόπωρο στο Πεκίνο θα μας δώσουν τη δυνατότητα να επιτύχουμε προόδο ε, στα κομμάτια που αφορούν τα κομμάτια της οικονομικής συμφωνίας που αφορούν θέματα ε, εμπορίου. Αυτό θα ενδυναμώσει και οικονομικά και πολιτικά τη σχέση μα. Κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου θα έχουμε διάφορε ευκαιρίε να συζητήσουμε την άρση των εμποδιών σε διμερέ επίπεδο ε, τομεακός διάλογος, ε, ε, η κοινή η επιτροπή στην οποία παρακαθίζουν μέλη της εκπρόσωπη της Ένωσης και της Κίνας. Αυτά θα μας δώσουν τη δυνατότητα να συζητήσουμε, αν όχι να επιλύσουμε τα προβλήματα που οδηγούν σε τριβές για να μην πω προς τριβές με την Κίνα, η οποία βεβαίως καλείται να σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις στα πλαίσια του ΠΟΕ όπως συμφωνίες για πρόσβαση στην αγορά, για τους παρόχους υπηρεσιών, IPR, διαφάνεια των τεχνικών κανονισμών και ούτω καθ' εξής. Η στρατηγική της Λισαβόνας είναι το βασικό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας για να αναπτύξουμε περαιτέρω την φορό ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Η ευημερία στην Ένωση βασίζεται εκ παραδόσεως στην εμπορική ευρωστία και την οικονομική βεβαίως ευρωστία των ευρωπαϊκών χωρών. Αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας πλέον με πιο λυρητό τρόπο. Ε, η πρωτοβουλία Global Europe του 2006 ήταν ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση για να δημιουργήσουμε αυτή τη συνολική στρατηγική σύμφωνα με την οποία το εμπόριο θα μπορέσει να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να συνεισφέρει στην διέξοδο ε, από την κρίση. Πρέπει να συνεχίσουμε να οικοδομούμε από αυτής της ε, βάσης και στα πλαίσια αυτά χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη κανονιστική συνεργασία σε σχέση με τις τρίτες χώρες. Το εξωτερικό εμπόριο και το άνοιγμα επίσης θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης όπως και όλα τα άλλα κομμάτια της στρατηγικής της Λισαβόνας. Δύο λόγια τώρα για τις διαπραγματεύσεις άκτα. Η Προεδρία έχει επίγνωση των διαφόρων, των πολυάριθμων ε, θεμάτων που θα πρέπει να επιλύσει το Συμβούλιο και των ερωτημάτων που έθεσε ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Συμβούλιο. Η Τσεχική Προεδρία μέσω του Υπουργού Ράιμαν έχει δώσει κάποιες απαντήσεις ήδη η πειρατεία, η παραποίηση των αυθεντικών προϊόντων, η συστηματική καταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων είναι τα βασικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στους αγορές των τρίτων χωρών. Στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και πολλές φορές θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια την ζωή ή την υγεία των καταναλωτών παγκοσμίω. Γι' αυτού του λόγου ε, υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία διαπραγμάτευση μια νέα εμπορική συμφωνία που θα βασίζεται στην ε, εφαρμογή τη συμφωνία ε, κατά τη παραποίηση των προϊόντων. Και θέλουμε να συνεισφέρουμε στην αναζωογόνηση των συζητήσεων αυτών, ούτω ώστε οι διαπραγματεύσει ενδεχομένω να ολοκληρωθούν επιτυχώ το 2010. Έχουμε την ίδια κατανόηση, την ίδια θεώρηση πραγμάτων και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσουμε τη σημαντική δουλειά που έχουμε να κάνουμε από ε, αυτού του θέματος ε, ξεχωριστά με κάθε εταίρο με τον οποίο διαπραγματευόμαστε για να επιτύχουμε τους στόχους της χιλιετίας. Όλοι οι τομείς, όλες οι πολιτικές μπορούν και πρέπει να ε, συνεισφέρουν στον ε, συνολικό στόχο της ε, εξαφάνισης της ένδυας, της φτώχειας στον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό εργαλείο και για τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και πιστεύουμε ότι οι πολιτικές αυτές, τα PCD δηλαδή, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να ε, δώσουμε νέα όθηση στις ε, επί της συζητήσεις που θα πρέπει να λάβουν χώρα. Επίσης, τα PCDA μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ χρήσιμο μέσο για, την, ε, για τον καθορισμό μιας εμπορικής πολιτικής της Ένωσης που θα πρέπει να είναι ακόμα πιο φιλική προς το περιβάλλον από ό,τι είναι σήμερα. 16 με 17 Νοεμβρίου θα εγκρίνουμε συμπεράσματα του Συμβουλίου για το μελλοντικό σχεδιασμό της διαδικασία PCD και είναι πολύ σημαντικό η διαδικασία PCD να συμπεριλαμβάνει και επιχειρησιακές προτάσεις, πρακτικές προτάσεις που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να αναπτύξουμε συγκεκριμένες στρατηγικές. Θα πρέπει να επικεντρώσουμε δε την προσοχή μας στις προτεραιότητες που αποτελούν την κύρια μέρημνα των αναπτυσσομένων χωρών. Για τη δική μας εμπορική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις μελέτες αντικτύπου για το πώς το εμπόριο πλήττει, του στοχ... Ε, επηρεάζει τους στοχούς ε, ανά τον κόσμο. Ας περάσω τώρα στο εμπόριο και το κλίμα. Η καταπολέμηση της αλλαγής ε, του κλίματος είναι πρώτη στην προτεραιότητα για την Προεδρία μας και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη στην Κοπενχάγη τον Δεκέμβριο ε, μιας αφιλόδοξης συμφωνίας. Η διάσκεψη αυτή θα είναι κρίσιμη για να μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα υπέρ του κλίματος. Αυτό θα αποτελέσει σημαντική πρόκληση. Θα χρειαστεί όλοι οι συμβαλόμενοι να συμβάλλουν με τρόπο επικοδομητικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει ηγετική, ηγετικό ρόλο, να παίξει ηγετικό ρόλο. Τα θέματα <clears throat> εμπορίου δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμω ότι δεν πρέπει για τα θέματα αυτά να δραστηριοποιούμαστε σε, από άλλων βημάτων. Πρέπει να συμβάλλουμε στη συνολική προσπάθεια για τη μετρίαση των δυσμενών συνεπειών της αλλαγής του κλίματος. Είμαι πεπισμένοι ότι για να προχωρήσουμε επικοδομητικά χρειάζεται να βρούμε τρόπου να χρησιμοποιήσουμε ρυθμίσεις του εμπορίου και των αγορών για να ε, βελτιώσουμε το περιβάλλον. Να κάνουμε και πρόοδο στις ε, συζητήσεις DDA για να ε, καταργήσουμε όλους τους φραγμούς και τους δασμούς στο εμπόριο και στις υπηρεσίες που έχουν σχέση με το περιβάλλον. Αυτό θα βελτιώσει την κατάσταση του κλίματος χωρίς ταυτόχρονα να επιδεινώσει την οικονομική κατάσταση. Χρειάζεται να επεξεργαστούμε και τις προδιαγραφές την ε, επισήμανση διετικετών ε, των διαφόρων προϊόντων κλπ. Που έτσι και με τον τρόπο αυτό θα διευκολύνουμε το εμπόριο. Ιδιαίτερα να αποφύγουμε οι προδιαγραφές αυτές να γίνουν νέα εμπόδια, νέα κολλήματα για τις εξαγωγές. Το, ο Οργανισμός Πιστοποίησεως θα κάνει μια σχετική διάσκεψη στη Στοκχόλμη τέλη Νοεμβρίου. Η προώθηση της κοινωνικής ευθύνης των εταιριών είναι επίσης σημαντικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε, σε, σε άλλους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην αηφόρο ανάπτυξη καθώς και στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Εν προκειμένου μπορώ να ανακοινώσω ότι στη διάρκεια της Προεδρίας μας θα διεξαγάγουμε σχετική διάσκεψη στις 11 και 12 Νοεμβρίου στη Στοκχόλμη με θέμα προστασία, σεβασμός και ε, μέσα αποκατάστασης. Λίγα λόγια ακόμα σχετικά με τις άλλες προκλήσεις της, ε, που αντιμετωπίζει η εμπορική πολιτική και επί του παρόντος αλλά και στο μέλλον. Στην ε, ε Σουηδική Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον έγινε πριν από λίγο καιρό μια συνάντηση για να συζητηθούν σχετικά θέματα. Οι ροές του διεθνού εμπορίου και ε, ε, επενδύσεων έχουν αλλάξει. Το εμπόριο διεξάγεται τώρα μεταξύ διαφόρων μονάδων πολυεθνικών επιχειρήσεων, διότι αυτό υπαγορεύουν οι εξελίξεις ε, στις ροέ. Και ταυτόχρονα οι διαπραγματεύσει γίνονται ακόμα με καθαρά εθνικά, εθνικά κριτήρια. Και γίνονται όλο και πιο σημαντικά άλλα εμπόδια εκτός από τους παραδοσιακούς δασμούς. Οι εμπορικές πολιτικές πρέπει να αντιμετωπίσουν λοιπόν σημαντικές προκλήσεις όπως και του κλίματος και της ανάπτυξης. Στη διάρκεια της Προεδρίας μας θα συνεχίσουμε τη σημαντική αυτή συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συζήτηση η οποία θα συμβάλλει και στον θετικό ρόλο ε, που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο, ε, στη Γενέβη, στην Υπουργική Διάσκεψη. είμαστε άντρες και γυναίκες πολιτικοί που ασχολούμαστε με το εμπόριο. Ωστόσο, η παγκόσμια οικονομία είναι παγκόσμια και η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι να προσαρμοστεί η εμπορική πολιτική στις κοινωνίες και στους καιρούς μας. Και εσείς ως μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου έχετε ιδιαίτερο ρόλο που ε, καλείστε να παίξετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε και να συμβάλλετε αλλά και να αμφισβητήσετε τι εμπορικέ μα πολιτικέ. Η δική σα συμβολή λοιπόν είναι ουσιώδε τμήμα τη συνολική προσπάθεια τη Ένωση να αναπτύξει την εμπορική πολιτική. Μαζί εσεί και εμεί μπορούμε να εξηγήσουμε και στου πολίτε μα, αλλά και στου εταίρου μα τα ωφελήματα που απορρέουν από το ελεύθερο εμβόλιο και τι ανοιχτέ αγορέ. Αναμένω να συνεργαστώ μαζί σα σε πνεύμα ανοιχτό. Ολοκληρώνω εδώ. σα ευχαριστώ που παρακολουθήσατε με προσοχή την μακρά μου ομιλία και αναμένω να ακούσω και τις δικές σας απόψεις ή και να απαντήσω στις ερωτήσεις, μας, στις ερωτήσεις σας. Thank Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Ίσως ήταν λίγο συντομότερος ο λόγος σας από ό,τι είπατε στην αρχή, πάντως ήταν ιδιαίτερα περιεκτικός και σε πολλά σημεία ανταποκριθήκατε στις προσδοκίες των συναδέλφων. Άκουσα με ενδιαφέρον τις διμερείς συμφωνίες και συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Και θα κάνω και ε, ερωτήσεις, αλλά πρώτα δώσουμε το λόγο στον Δανιέλ Κάσπαρη του Λαϊκού Κόμματος. Ε, συντονιστές θα λάβουν το λόγο με τη σειρά. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ που προσήλθατε εδώ και εξ ονόματο τη ομάδα του κόμματό μου. σα εύχομαι και σε εσά και στην κυβέρνησή σα επιτυχή Προεδρία. Λίγα σχόλια για τα όσα είπατε. Αφενός, όταν μιλείτε για τον ΠΟΕ και την ένταξη τη Ρωσία στον οργανισμό αυτό, νομίζω ότι με την υποδοχή τη Ουκρανία δεχθήκαμε ορισμένε εξαιρέσει ω Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν θα πρέπει ωστόσο να δεχθούμε σε καμία περίπτωση στην περίπτωση τη Ρωσία για παράδειγμα για την ενέργεια ή για ορισμένα είδη Θα ήθελα πολύ να ακούσω την θέση σας και κυρίως να μείνετε, ε, μείνετε στη θέση αυτή. Τώρα για, την, ε, για τις εμπορικές με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η διατλαντική αγορά για την δική μας ευρωπαϊκή οικονομία έχει ιδιαίτερη σημασία. Θα, θα ήθελα να θίξετε με τους Αμερικανούς εταίρους θέματα ιδίω εκείνων των πολιτικών όπου μπορούμε να επιτύχουμε. Μέχρι τώρα έχουμε συζητήσει ιδίω για θέματα όπου υπήρχαν προβλήματα, όπως Airbus και Boeing, όπως διάφορα άλλα θέματα όπου είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες μαζί τους. Θα ήθελα πολύ τώρα να ρίξετε ιδιαίτερο βάρος, να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα εκείνα όπου μπορούμε με τους Αμερικανούς να επιτύχουμε πάρα πολλά. Μιλούμε για ένα όγκο συναλλαγών της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας επιθυμείτε να ολοκληρώσετε δύο εμπορικές συμφωνίες, υποθέτω ότι εννοείται με την Νότια Κορέα και με τον Καναδά. Θα χαρούμε πάρα πολύ να προχωρήσετε σε αυτό. Προωθήσετε ωστόσο και συμφωνία με την Ινδία. Και εάν δεν καρποφορήσει η προσπάθεια αυτή ακόμα στη δική σας Προεδρία, τότε ελπίζω στην επόμενη. Ε, είπατε επίσης ότι θα θέλατε η εμπορική πολιτική να μπορεί ε, να στηρίζει και τους στόχους της Κομπεχάγης. Εγώ συμφωνώ, γιατί μπορεί η εμπορική πολιτική να υποστηρίξει και πολλά θέματα της ε, πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, με εξαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας, με σχετικές συνεργασίες. Αλλά εξακολουθούμε να μιλούμε για αμυντικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ δεν μιλούμε για border tax adjustment ποια μπορεί να είναι η συμβολή θετικών μέτρων, εκτός των αμυντικών μέτρων. Και τελικά το αποτέλεσμα των αμυντικών μέτρων που λαμβάνουμε, ποιο είναι. Κάτι που δεν άκουσα ήταν σχετικά με την ε, στρατηγική των πρώτων υλών. Πέρσι εγκρίναμε και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμα τη στρατηγική για τις πρώτες ύλες. Έχουμε ωστόσο λάβει αυτές τι αποφάσεις. Αφού τις λάβαμε, θα πρέπει τώρα να φροντίσουμε να μην απολέσουμε από το πτικό μας πεδίο το θέμα των πρωτονυλών. Ναι, μεν έχει χαλαρώσει και μάλιστα με δραστικότατο τρόπο η κατάσταση στο, στο παγκόσμιο επίπεδο για τις πρώτες αλλά μην γελιέστε, οι Κινέζοι προωθούν την πολιτική τους αγοράς παντός είδους πρώτων υλών με ρυθμούς. Κατά τα άλλα, εξακολουθούν να, έχουν, να ακούγονται ορισμένε ιδέε οι οποίε δεν είναι σωστέ. Για παράδειγμα, για την προστασία βιομηχανική ιδιοκτησία. Που ε, ορισμένε από τι ιδέε αυτέ ανοίγουν και τι ε, ε πόρτε για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Θα ήθελα πολύ να επανέλθετε και σε αυτό και κυρίως να τηρήσετε τι ε, θέσεις που είπατε. Και τέλο, μιλήσατε και για κολλήματα στις συναλλαγές μη δασμολογικού χαρακτήρα. Θυμίζω εν προκειμένου αντιτρομοκρατικά μέτρα. Για παράδειγμα, την σάρωση ε, εμπορευματοκιβωτίων στις Ηνωμένες Πολιτείες στα σημεία εισαγωγής τους στη χώρα αυτή. Θα ήθελα να παρακαλέσω να φροντίσετε και στο θέμα αυτό ώστε παρά τις ανάγκες βέβαια της ασφάλειας, τα μέτρα, τα αντιτρομοκρατικά αυτά μέτρα να μην γίνουν εν τέλει στην πραγματικότητα εμπόδια στις εξαγωγές. Σας ευχαριστώ και πάλι και σας εύχομαι καλή επιτυχία στις προσπάθειές σας. Ας ακούσουμε τρεις ερωτώντες Έναν ακόμη λοιπόν ε, συντονιστή. Κύριε Ρίφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Υπουργέ για τα όσα ακούσαμε. Εκ μέρους της ομάδας μου θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας τους επόμενους μήνες. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον όλα τα όσα είπατε και υπάρχουν θέματα στα οποία θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Ένα ερώτημα γενικό καταρχάς που για εμάς αποτελεί προτεραιότητα, για εμάς ως πολιτική ομάδα, αλλά και για την Κομισιόν θεωρώ, που έχει να κάνει με την ε, ενίσχυση της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η άποψη των ε, εκλεγμένων αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εμπορική πολιτική. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω την άποψή σας για αυτό, πώς σκοπεύετε θεσμικά να ενισχύσετε το ρόλο της Επιτροπής ΙΝΤΑ και πώς θα ενισχύσετε τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, γιατί είναι αλήθεια ότι σε αυτό το τομέα το τόσο σημαντικό του διεθνούς εμπορίου θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παραμεριστεί σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο παρόλο που κάποια θέματα δεν είναι τόσο εύκολα ούτε να τα εγκρίνουμε, ούτε να τα εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας. Τώρα, όσον αφορά τις ε, τρέχουσες διαπραγματεύσεις. Στην προηγούμενη θητεία είχαμε ασχοληθεί με τη ζώνη Euromed και είχε φανεί ότι θα ήταν δύνατο να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις πριν το 2010. Υπάρχουν ε, περισσότερες πληροφορίες που θα μπορούσατε να μας δώσετε τώρα για αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ε, έχει δίκιο ο κύριος Κάσπαρη για το θέμα της Κορέας. Συζητήσαμε χτες το θέμα με τον Γενικό Διευθυντή της ε, Επιτροπής. Πάντως, μία συμφωνία με την Νότια Κορέα, ειδικά στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, είναι σημαντική, όμως υπάρχουν και πολλές επιφυλάξεις και φόβοι. Και θα έπρεπε να δούμε τι θα γίνει με το θέμα της πρόσβασης ε, που θα έχουμε εμείς, αλλά και τους φόβους που υπάρχουν για πιθανή εισβολή των κορεατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Όσον αφορά τις EPA, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί εμάς και τους συναδέλφους τους τελευταίους μήνες. Έχουμε την ε, εντύπωση ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση δεν έχει προχωρήσει όσο θα έπρεπε. Γνωρίζουμε βεβαίως τις δυσκολίες που υπάρχουν σε πολλές ε, ζώνες ε, στην Αφρικανική Ήπειρο θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την άποψή σας και ειδικά για το θέμα ότι πολλές χώρες ΑΚΕ πλέον αρνούνται τις συμφωνίες, ειδικά χώρες όπως η Σιγκαπούρη που είναι και από τις πλέον ευνοευμένες. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις ανησυχίες της ομάδας μου και βεβαίως θα ακούσετε και άλλα σχόλια στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Καζάκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω και εγώ για την παρέμβασή σας και για τις ε, πολλές πληροφορίες που λάβαμε από εσάς, καθώς και για τις σαφείς σας δεσμεύσεις. Ως ε, μέλος της φιλελεύθερης ομάδας, ε, συμφωνώ απολύτως μαζί σας στο θέμα της αντιμετώπισης του προστατευτισμού. Θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, ειδικά στα πλαίσια της σημερινής οικονομικής ύφεσης. Είμαστε πεπισμένοι ότι το εμπόριο είναι η εμπροστοφυλακή της ε, οικονομικής ανάκαμψης που θα βοηθήσει στην ε, ανάκαμψη της ανάπτυξης ε, και της ε, απασχόλησης. Οπότε, το θέμα των ε, μη δασμολογικών εμποδίων είναι πολύ σημαντικό πλέον, γιατί πρέπει να έχουμε όλη ίση πρόσβαση στις παγκοσμίες αγορές. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω και τι ακριβώς αναμένετε από τον νέο της Ντόχα Σήμερα το πρωί είχαμε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων με τον πρέσβη της Κίνας για τα προβλήματα που προέρχονται από την Κίνα και αφορούν τις ευρωπαϊκές εξαγωγές, ειδικά όσον αφορά τα μη δασμολογικά εμπόδια και προβλήματα. Και επίσης συμφωνήσατε, σημειώσατε μάλλον, το ρόλο της Ρωσίας και την πιθανότητα ένταξης στον ΠΟΕ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ειδικά όσον αφορά τις ενισχύσεις για την εξαγωγή ρωσικής ξυλίας, αν ε, έχετε καταλήξει σε μία αποδοχτή λύση. Ένα άλλο θέμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι αυτό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η άποψή σας είναι καινοτόμος ε, και νομίζω ότι θα έπρεπε να αντιλάβουν υπόψη της όλοι οι οικονομικοί παράγοντες ε, των ευρωπαϊκών κρατών. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε πρώτα τους πέντε συντονιστές και μετά τις ερωτήσεις των υπόλοιπων μελών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Είναι επίσης ενδιαφέρουσα η σύνδεση της δικής σας παρουσίασης με την παρουσίαση του κυρίου Οσάλιβαν χτες προκύπτουν διάφορα πολιτικής φύσης ε, θέματα που έχουν να κάνουν και με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με τα κοινωνικά θέματα. Ο κύριος Σάλιβαν μας είπε ότι όλα αυτά δεν είναι δική του αρμοδιότητα, αλλά αρμοδιότητα του Συμβουλίου. Και το Συμβούλιο είναι αυτό που θα έπρεπε να εξελίξει κατάλληλα τις αρμοδιότητες της Επιτροπής σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω κάποιες διευκρινήσεις για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και θα ήθελα να ακούσω ποιος νομίζετε ότι θα έπρεπε να είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της Ονδούρας, αν σκοπεύετε να καταργήσετε το προτιμησιακά καθεστώς, αν πρόκειται να συνεχίσετε τις σχέσεις ε, με την κυβέρνηση της Ονδούρες, ε, ακόμη και σε θέματα που έχουν να κάνουν με τεχνικές συμφωνίες. Επίσης, κυρία Υπουργέ, αναφερθήκατε στην ολοκλήρωση του γύρου της Ντόχας. Μήπως μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι απόψεις σας ε, για τις νέες θέσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης. Να μας πείτε επίσης αν είχατε επαφές με την κυβέρνηση Ομπάμα, τον ΙΠΑ και αν ε, βλέπετε με αισιοδοξία το μέλλον όσον αφορά τη συμμετοχή της Αμερικής σε αυτό το γύρο ή αν θα πρέπει να συνεχίσει να καθοδηγεί τις εξελίξεις μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ. Αναφερθήκατε και στη διάσκεψη της Κοπενχάγης. Στο τέλος ε, του εξαμήνου η Προεδρία σας ε, θα έχει την ε, δυνατότητα τόσο στη Γενέβη όσο και στη διάσκεψη της Κοπενχάγης να παίξει σημαντικό ρόλο. Επειδή είπατε ότι το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας θα είναι σημαντικό για τη διάσκεψη της Κοπενχάγης και επειδή κατά αυτόν τον τρόπο έτσι θα ολοκληρωθούν οι συζητήσεις στα πλαίσια του ΠΟΕ για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, θα ήθελα να πω ότι γνωρίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις ε, της Ντόχας εξακολουθούν για πολύ καιρό. Από την άλλη πλευρά, το θέμα της διάσκεψης της Κομπεχάγης είναι σαφώς πιο επίγον και θα ήθελα να μάθω πώς εντάσσεται στο εμπορικό τομέα. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω τι πρωτοβουλία σκοπεύει να πάρει η Σουηδική Προεδρία προκειμένου προληπτικά αν θέλετε να προκύψει ε, μια κατά κάποιο τρόπο ελάφρυνση του όλου θέματος της πνευματικής ιδιοκτησίας ε, στην Κομπεχάγη. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι ο τελευταίος συντονιστής και θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος. Καταρχάς σας ευχαριστώ για την ειλικρίνειά σας. Άκουσα αυτά που είπατε για τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Εγώ πάντα ήμουν υπέρ των πολυμερών συμφωνιών στα πλαίσια του ΠΟΕ, αλλά πλέον βλέπουμε ότι συχνά καταλήγουμε στις διμερείς διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω αν μετά τον Οκτώβριο του 2008 υπήρξαν επιπλέον διαπραγματεύσεις με την Λιβύη και αν είμαστε πλέον υπέρ μια συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τη Λιβύη. Το ίδιο ισχύει και για το Πακιστάν. Γνωρίζω ότι η Βρετανία ενθαρρύνει ιδιαίτερα την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Πακιστάν. Μετά και από την ε, διάσκεψη κορυφής φέτος. Και από ό,τι φαίνεται αυτό το ενθαρρύνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Συμβούλιο λοιπόν θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα μια τέτοια συμφωνία με το Πακιστάν, η ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Ας ξεκινήσω από την αρχή. Το πρώτο θέμα ήταν ε, η σχέση εμπορικής πολιτικής, Κοπενχάγη, θέματα που έχουν να κάνουν με το κλίμα και το πώς συνδέονται με το εμπόριο. Πώς θα εντάξουμε το εμπόριο σε αυτά τα θέματα. Πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εμπορική πολιτική ως θετικό εργαλείο στα πλαίσια της αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ανησυχίες και τα συμφέροντα των αναπτυσσόμενων χωρών, βεβαίως. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε μια θετική ατζέντα, να αναφέρουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες σε θέματα που θα έχουν να κάνουν με την εξαγωγή προϊόντων και τεχνολογιών πιο φιλικών προς το περιβάλλον και την δημιουργία και τέτοιων υπηρεσιών σε αυτές τις χώρες. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε θετικές εξελίξεις στο άμεσο μέλλον εδώ. Επιπλέον, θα πρέπει να ασχοληθούμε με τον στόχο της επίτευξης διεθνών λύσεων που θα ενισχύουν τις πρωτοβουλίες μας ε, στον τομέα του κλίματος. Και παράλληλα με τα πρότυπα που υπάρχουν για την μείωση των εκπομπών. Βεβαίως, η ύπαρξη κλιματικών προτύπων για την μείωση των εκπομπών αερίου, αερίων του θερμοκηπίου, πρέπει να συνδυαστεί με μια προσπάθεια για τη μη δημιουργία εποδίων στο εμπόριο, ειδικά για τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό θα το συζητήσουμε στη Στοκχόλμη 23 με 25 Νοεμβρίου. Η συζήτηση είχε ξεκινήσει ήδη από το Δεκέμβριο του 2007 στη διάσκεψη του Μπαλί είχαμε συζητήσει το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπορική συνεργασία για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Παρόλα αυτά, να πω ότι αυτή τη φορά στη διάσκεψη της Κοπενχάγης οι κλιματικές αλλαγές δεν θα αποτελέσουν τμήμα της συζήτησης. Τώρα, στο θέμα της στρατηγικής μας μετά την κρίση. Συμφωνώ ότι είναι σημαντικό το θέμα. Στην ομιλία μου σας μίλησα για την Ρωσία και για το θέμα των δασμών για την εξαγωγή. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι αυτό της Ουκρανίας ε, και της ενέργειας. Επίσης, ε, η GCC και η εξαγωγική. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε αυτή τη στρατηγική μας. Το θέμα αφορά και την Κίνα. Υπάρχουν πολλά θέματα που προκύπτουν όσον αφορά την πρόσβασή μας σε πρώτες ύλες. Και Όσον αφορά τα NTB, αυτό που μπορώ να πω από σουηδικής πλευράς είναι ότι είχαμε μια διασκέψη φέτος στην Άνοιξη και ρωτήσαμε εταιρείε ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που θα θέλατε για να αυξήσετε την εμπορική σας δραστηριότητα. Οι περισσότεροι απάντησαν ολοκλήρωση του γύρου της Ντόχα και η δεύτερη προτεραιότητα ήταν τα NTBs ή τα μη δασμολογικά εμπόδια δηλαδή και τα εμπόδια τέτοιου είδους που αντιμετωπίζουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνας τώρα, και το πώς επηρεάζει την Επιτροπή Ίντα. Έλαβα υπόψη μου την άποψη της ίντα όπως ε, αναφέρθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου από το Μάιο. Όπως γνωρίζετε, δεν έχει ακόμη επικυρωθεί η συνθήκη της Λισαβόνας από όλα τα κράτη-μέλη. Στις 2 Οκτωβρίου θα έχουμε το νέο δημοψήφισμα στην Ιρλανδία και αν το αποτέλεσμα είναι ευνοϊκό για τη συνθήκη, η Σουηδία θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να μπορέσει να τεθεί άμεσα σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε την καλή συνεργασία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και από τη στιγμή που θα τεστηθεί σε ισχύ η συνθήκη. Η νέα συνθήκη αυξάνει τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου σε πολλούς τομείς. Η Προεδρία θα ήθελε να έχει διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την εφαρμογή της νέας συνθήκης. Τώρα, για τις συγκεκριμένες συνέπειες της συνθήκης δεν θα ήθελα να περάσω τώρα σε λεπτομέρειες ή να κάνω προβλέψεις. Θα προτιμούσα να μπούμε σε λεπτομέρειες αφού τεθεί σε ισχύ η συνθήκη. Αφού λοιπόν δούμε τα αποτελέσματα της Δευτέρας Οκτωβρίου. Ένα άλλο ερώτημα αφορούσε το Euromed και το ποιες θα είναι οι εξελίξεις εκεί. Δεν είμαι σίγουρη αν σας άκουσα καλά, αλλά με ρωτήσατε μάλλον αν θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις το 2010. Δεν ήμουν σίγουρη αν άκουσα αυτό. Μετά την κατάσταση στη Γάζα είχαμε πάγωμα των ε, συναντήσεων, κάτι που δημιούργησε προβλήματα. Βεβαίως θεωρούμε ότι κάποιες διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους. Εν πάση περιπτώσει, η Προεδρία χαίρεται και επικροτεί το γεγονός ότι θα υπάρξει επανέναρξη των συναντήσεων και θα υπάρξουν τέτοιες συναντήσεις στο φθινόπωρο, αν και δεν έχουμε ακόμη επιβεβαιώσει ημερομηνίε. Um, about... Uh, Κατόπιν, Νότια Κορέα, αναφέρθηκε ένα σχετικό ερώτημα και αυτοκινητοβιομηχανία. Πώς βλέπουμε τα πράγματα στον τομέα αυτό. Είπα και προηγουμένως ότι η Κορέα είναι η τέταρτη μεγαλύτερη χώρα σε ό,τι αφορά τις εμπορικές ανταλλαγές. Μεταξύ 2003 και 2007 δε είχε ρυθμούς ανάπτυξης 10%. Οπότε ένα γενικό FTA με την Κορέα θα είναι πολύ σημαντικό βήμα πρόοδου και για το δικό μας και τη δικιά μας ατζέντα αλλά και εις ό,τι αφορά τη σύνοψη άλλων συμφωνιών FTA. Έχουμε εκτιμήσει ότι οι επιχειρήσεις μας ε, έχουν πολλά να κερδίσουν από μια συμφωνία ελευθερών με την ε, Κορέα. και να αυξήσουμε τις αγωγές μας στην Κορέα κατά 5,8% αυτές είναι εκτιμήσεις ε, που έχουμε κάνει. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ σημαντική δοκιμασία που θα αποδείξει αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προχωρήσει ή όχι. Σε ορισμένα θέματα εμπορικής πολιτικής. Όλοι βγαίνουν κερδισμένοι από τη σύναψη μιας συμφωνίας ελευθερού με την Κορέα. Δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ίδια η Κορέα. Τώρα, για την αυτοκινητοβιομηχανία, για την οποία έχουν εκφραστεί φόβοι ότι θα πληγεί με τη σύναψη μιας ενδεχόμενης συμφωνίας FTA με την Κορέα. Δεν αληθεύει κάτι τέτοιο. γιατί υπάρχει μια μεταβατική περίοδος 6,5 ετών. που μάλιστα έχει και κάποιες ρήτρες σταδιακής εφαρμογής. Οπότε δεν θεωρώ ότι φταθούν οι ανησυχίες και οι φόβοι για την αυτοκίνητο Προσωπικά δε, ως πολιτικός και ως Σουηδή, γιατί και εμείς έχουμε ε, δύο αυτοκινητοβιομηχανίες για τις οποίες ανησυχούμε. Η ΣΑΜΠ απειλείται με απώλεια 4.700 θέσεων απασχόλησης. Και αυτό μας έχει κάνει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Θα πρέπει να προσανατολίσουμε την εταιρεία αυτή προς άλλους τομείς. Έχουμε ας πούμε αναπτύξει πολύ τις τεχνολογίες που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Θα πρέπει να επαναπροσανατολίσουμε απλώς λοιπόν την, ε, τις δραστηριότητες της εταιρείας αυτής σε άλλους καινοτόμου τομεί. Είναι ευκαιρία λοιπόν και όχι απειλή. Και δεν θα πρέπει να αποτελέσει η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με την Νότιο Κορέα συνώνυμο της μιας συμφωνίας για την αυτοκινητοβιομηχανία. Αναδιάρθρωση λοιπόν. Σε παγκόσμιο μάλλον στα επίπεδα. Και υπάρχει καιρός. 6,5 χρόνια. Εμείς στη Σουηδία έχουμε ήδη ξεκινήσει. Αφρική. συμφωνίες ΕΠΑ. Σιγκαπούρη. Το έχουμε συζητήσει και κατά παρελθόν το θέμα και εμείς στη Σουηδία αναγνωρίζουμε την υπέρξη του προβλήματος. Η διευκόλυνση του εμπορίου, επενδύσεις, ανταγωνισμός, δημόσιες προμήθειες, πνευματικά δικαιώματα είναι τα κεντρικά σημεία μιας στρατηγικής εμπορικής πολιτικής. Και όπου βεβαίως οι χώρες εκεί θα πρέπει να έχουν μια αυτοδυναμία, να μην βασίζονται σε βοήθεια μόνο. Ούτε εμείς μπορούμε να επιβάλλουμε αυτά τα θέματα στους εταίρους μας. Οι υπηρεσίες, τελεπικοινωνίες, οικοδομές πρέπει να προσελκύσουν οι χώρες αυτές επενδύσεις. Κάθε έκθεση που έχει δημοσιευτεί για τις σχετικές επενδύσεις συμπεραίνει ότι για να γίνει αυτό χρειάζεται ένα διαφανές και ασφαλές επενδυτικό κλίμα. Και οι ΕΠΑ μπορούν να το επιτύχουν αυτό. Ας πούμε στην ΕΠΑ με την Καραϊβική περιλαμβάνονται ήδη κάποια κεφάλαια για τις υπηρεσίες. Κατανοούμε όμως και τις ανησυχίες των ε, χωρών αυτών και γι' αυτό έχουμε πολλές φορές πιο ελαστική ε, στάση στις ε, διμερείς σχέσεις που έχουμε με κάθε μία από τις χώρες αυτές. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Εξαγωγικοί δασμοί και ρήτρα πλέον ευνοουμένου κράτους. Να αναφέρω εδώ μια απο τις χωρες αυτες υπαρχουν και αλλα θεματα εξαγωγικοι δασμη και ρητρα πλεον ευνοουμενου κρατους να αναφερω εδω μια εμπειρια που είχαμε εμείς στη Σουηδία. Την περασμένη άνοιξη καλέσαμε μια σειρά πρεσβευτών αφρικανικών χωρών για να συζητήσουμε ποια είναι τα βασικά προβλήματα που εκείνοι πιστεύουν ότι υπάρχουν. Κάθε χώρα έλεγε ε, υπό το δικό της οπτική ε, γωνία τα πράγματα, αλλά ο κοινό παρανομαστής ήταν οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Οι αφρικανικές χώρες πάντα θεωρούσαν επ' αυτού του θέματος ότι ήταν... Ε, υπεροπτική η ευρωπαϊκή πλευρά. Ότι δεν άκουγε τι είχαν να πούν οι Αφρικανοί. Μόλις το καταλάβαμε αυτό, αλλάξαμε το κλίμα των διαπραγματεύσεων. Χρειάζεται καιρός, χρειάζεται να μάθουμε, να ακούμε Χρειάζεται να μάθουμε να κατανοούμε τις ανησυχίες των χωρών αυτών. Then it was a question about uh, what... Κατόπιν. Ντόχα. Όπως είπα και στην ομιλία μου, η Ντόχα είναι οι τρεις πρώτες προτεραιότητες της Προεδρίας μας. Και θέλουμε βεβαίως ως βασική προτεραιότητα να περάσουμε το μήνυμα της ενότητος. Όλοι μαζί θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των διαπραγματεύσεων αυτών, διότι υπάρχουν πολλές χώρες που προσπαθούν να μας διαιρέσουν, να μας διχάσουν να αποσταθεροποιήσουν την κατάσταση. Εκπείρας, εφόσον έχουν καταρρεύσει οι διαπραγματεύσεις πολλές φορές, γνωρίζουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Ελπίζουμε όμως ότι θα αλλάξει το κλίμα. Πρέπει ένθεν και ένθεν να γίνουν περισσότερες παραχωρήσεις και εμείς από την πλευρά μας να κάνουμε χειρονομίες, αλλά και οι εταίροι μας ότι πρόκειται για αναπτυξιακό γύρο. Δηλαδή για τις αναπτυσσόμενες χώρες γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Με τις δηλώσεις ομάδας των 8, με τις δηλώσεις ομάδας των 20 για αποφυγή προστατευτισμού κτλ. κτλ. Νομίζω ότι έχουμε, τουλάχιστον εγώ έχω πλέον την πεποίθηση ότι θα προχωρήσουν τα πράγματα το φθινόπερο και σε τεχνικό και σε πολιτικό επίπεδο. Θα δούμε βεβαίω τι θα γίνει και στην Υπουργική διάσκεψη. Αλλά το 2010 θα πρέπει να είναι καταληκτική προθεσμία, διότι αλλιώς, αλλιώς όλοι θα βγούμε χαμένοι. Και ιδιαίτερα οι αναπτυσσόμενες χώρες. Okay. <laughs> okay. Mm. Eh, then... Eh, και μία ερώτηση για την ένταξη της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου καθώς και για τη ρωσική ξυλία. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι η Ρωσία πρέπει να πληρεί όλα τα κριτήρια όπως ισχύει για άλλες χώρες πριν να μπορέσει να ενταχθεί στον ΠΟΕ. Ένα από τα κριτήρια είναι βέβαια να μην προσθέσει και άλλους δασμούς στην ξυλία, αντίθετα να του μειώσει. Και μέχρι τώρα, από ό,τι φαίνεται, η προσπάθεια έχει αναβληθεί για ένα χρόνο. Πάντως θα προχωρήσουμε και το μήνυμα που λάβαμε την Άνοιξη είναι ότι θα συνεχίσουμε ότι θα συνεχιστούν οι συζητήσεις με τη Ρωσία για να δούμε πότε θα ε, μπορέσει η χώρα αυτή να ενταχθεί. και μια πιο συγκεκριμένη ε, συζήτηση για τη σχέση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ονδούρας. Τι θα γίνει τώρα μετά από το πραξικόπημα στην χώρα αυτή. Πάντως εγώ είμαι ικανοποιημένη που καταλήξαμε σε ένα συμβιβασμό μεταξύ των διαφόρων απόψεων στο Συμβούλιο. Έχουν οι διαπραγματεύσει για την ώρα ανασταλεί. Η ε, Προεδρία έχει τονίσει την ανάγκη να ε, ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσει όταν θα αποκατασταθεί η συνταγματική τάξη στην Ονδούρα. Και παρακολουθούμε προσεκτικά τις εξελίξεις στην χώρα αυτή η εξέλιξη είναι σημαντική και για την Ονδούρα αλλά και για όλη την περιοχή αυτή του κόσμου. Να μπορούμε να συνεχίσουμε με τις διαπραγματεύσεις δηλαδή το δυνατόν συντομότερο. Ακολουθεί η Λιβύη και το Πακιστάν. Σχετικά με την Λιβύη βρισκόμαστε στην αρχή των διαπραγματεύσεων. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος. Και πάντως μια μελλοντική FTA θα πρέπει ε, να ακολουθήσει μια ένταξη της χώρας αυτής στον ΠΟΕ. Σε ό,τι αφορά το Πακιστάν και τις ε, σχετικές συμφωνίες FTA έχουν προταθεί μέτρα από το Συμβούλιο για να τονωθούν οι εξαγωγές από το Πακιστάν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που κάτι που θα επιτρέψει στενότερη συνεργασία και που αυτή θα εξομαλύνει τον ε, δρόμο για μια μελλοντική FTA. Αλλά βέβαια δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ για τις πλήρες, πλήρες απαντήσεις. Εάν όλοι μιλήσουν σύντομα, πραγματικά ένα λεπτό δηλαδή, τότε ε, θα, μπορέσουμε να ακούσουμε και εσάς. Ο κύριος Ρινάλντι. think I, I just dropped. Αποσύρωμαι, Πρόεδρε. Ε, tack så mycket, herr ordförande. Ε, ja, det blir lite lustigt nu när... Ο κ. Χέλνερ. Ευχαριστώ. Είναι περίεργο που είχαμε πολύ χρόνο στην αρχή και πολύ περιορισμένο τώρα. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Με απασχολεί και εμένα ο προστατευτισμός στα πλαίσια της κρίσης. Το θέμα είναι, χρειαζόμαστε να χρειάζεται να δούμε κάποιον να ασκεί έναν ηγετικό ρόλο. Λέμε ότι δεν θέλουμε να, επιβάλλονται, να επιβληθούν νέοι ε, δασμοί και το καθεξής. Το βλέπουμε όμως από τις χώρες G20. Εμείς υποσχεθήκαμε ότι δεν θα επιβάλλουμε νέους φραγμούς, αλλά το βλέπουμε να γίνεται ξανά και ξανά. Και ε, αυτό θέτει ερωτήματα σχετικά με τις πολιτικές που ακολουθούνται για ε, την ενίσχυση της βιομηχανίας, για παράδειγμα, για ε, δασμούς που επιβάλλονται σε ρωσικά φορτηγά, που οι Ρώσοι ισχυρίζονται ότι είναι το ίδιο σαν να υποστηρίζουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία φορτηγών αυτοκινήτων. Μια τέτοια πολιτική δεν αποτελεί απειλή μονάχα τις μικρότερες αγορές, αλλά απειλεί και τις σχέσεις μας με άλλες χώρες. Και ένα θέμα ακόμη, αν με επιτρέπετε, που γνωρίζω ότι σας ενδιαφέρει και εσάς, μιλήσατε για το εμπόριο και, τις, και την κλιματική αλλαγή. Και είναι σωστό να είναι μηδενική η φραγμή, η δασμή, συγγνώμη. Και είπατε ότι μέσα στον γύρο της τόχα, θα ε, υπάρχει τάση και θα γίνει προσπάθεια να είναι μηδενική η φραγμή για ή δασμοί συγγνώμη και πάλι, για ε, προϊόντα τα οποία είναι περιβαλλοντικής ε, τεχνολογίας. Ε, θα ήθελα να ακούσω την άποψη σας. Κυρία Λούκας, τρεις σύντομε ερωτήσεις. Μιλάω γρήγορα όμως. Πρώτον, ήμουν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και δεν άκουσα την παρουσίασή σας Εκεί ε, συζήτησα θέματα παράνομης ξύλευσης στην ε, παράνομη συλλοτομία με τον ε, συνάδελφό σας. Θα υπάρξει συμφωνία. Όταν θα υπάρξει αυτή η συμφωνία θα θέσετε το θέμα της παράνομης υλοτομίας στην Ινδονησία και θα ασκήσετε πίεση για να σεβαστούν τα, τις συμφωνίες που ισχύουν γιατί, γιατί η παράνομη υλοτομία έχει βαρύτερα συνέπειε και στο περιβάλλον και έχουμε και την Κομεχάγη που επίκειται. Εξάλλου, ο κ. Σάλιβαν είπε ότι ε, προχωρούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά για το ε, Συμβούλιο που θεωρεί ότι ε, συμφωνία με την Κολομβία για την ώρα δεν είναι καλή ιδέα γιατί υπάρχει πραγματική δίωξη των συνδικαλιστών στην Κολομβία. Ελπίζω ότι οι πολιτικοί και στο Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο θα συμφωνήσουν ότι πρέπει να ανασταλούν οι συμφωνίες με την Κολομβία για να καταστεί σαφές στις αρχές αυτές ότι δεν θα ρινουμε μια τέτοια στάση. Πρόεδρε, στρέφομαι σε εσά για να πω ότι δεν είναι δυνατόν στην Επιτροπή, στη συνεδρίαση της Επιτροπής, να δίδεται ένα λεπτό ομιλίας. Στην Ολομέλεια, ναι, το καταλαβαίνω. Ένα λεπτό της ώρας. Λοιπόν, αποσύρωμαι κι εγώ ε, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, Πρόεδρε. Um, Peter. Thank you, Chairman. Σάστινη, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Πρώτα, ε, καλωσορίζω και συγχαίρω την κύριε Υπουργό, νομίζω θα απέκτησε πολλούς φίλους εδώ στην ε, Επιτροπή Ίντα με την πλήρη και ενδιαφέρουσα παρουσίασή της και έβαλε και τις DDA στην τρίτη ε, νομίζω ε, προτεραιότητα το ίδιο για τις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις και εγώ είμαι ιδιαίτερα ένθερμος οπαδός του Καναδά και πολύ ωραία τα είπε αλλά είπε λίγα για την Νότια Κορέα αν μπορεί να προσθέσει κάτι Εγώ έθιξα το θέμα χθε στην συζήτηση με τον κύριο Οσάλιβαν. Εξετάζοντα και τι δύο πλευρές, βλέπω και κατά τη γνώμη μου ότι η βιομηχανία γίνεται στην ουσία ο αποδιοπομένο τράγο στην ε, ε, συμφωνία FTA με την Κορέα. Μας είπαν χθε ότι είναι το θέμα των δασμών που θα μειωθούν σταδιακά μέσα σε 6,5 χρόνια, αλλά είχαν, τους είχαν υποσχεθεί ε, μια, ε, μια μελέτη ε, επιπτώσεων, την safeguard Plus Δεν έγιναν τα πράγματα αυτά. Και με τους νέους δασμούς και με, τις νέες, και με τα νέα κολλήματα των εξαγών που δεν είναι δασμοί, δεν βλέπω να έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Εσείς που είστε Σουηδοί και η Σκάνια είναι μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία. Εγώ είμαι Σλοβάκος, αλλά η αυτοκινητοβιομηχανία είναι μεγάλη υπόθεση για την Ευρώπη. Μπορείτε να προσθέσετε κάτι σχετικά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εσά κυρία Υπουργέ. Για την αυτοκινητοβιομηχανία με ερώτηση. Μια ερώτηση. Είπατε ότι στη Σουηδία η αυτοκινητοβιομηχανία θα πρέπει είτε να ε, αναδιαρθρωθεί ενδεχομένω και να ε, πάψει να λειτουργεί. Αυτό σημαίνει ειδικά για τη Σουηδία. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποιο νόημα η προμήθεια αυτοκινήτων στην Ευρώπη, με αυτοκίνητα κατασκευασμένα στην Ευρώπη, ε, να μην έχει νόημα. Θα ήθελα να κάνετε μια διευκρίνηση. Θα προσπαθήσω να είμαι ε, σύντομη. Δύο ερωτήσεις που δεν απάντησα πριν. Πρώτα, τι πιστεύω σχετικά με τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση. Είναι σημαντική η ερώτηση αυτή. Είναι σημαντικό για μας να συνεργαστούμε μαζί τους, να επιτύχουμε τη συνεργασία τους, γιατί αλλιώς ούτε στον γύρο της Ντόχα, ούτε αλλού θα μπορέσουμε να επιτύχουμε περισσότερη συνεργασία με ταξί Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι επίσης σημαντικό να συζητήσουμε ε, και τα θέματα του Διατρατικού Οικονομικού Συμβουλίου. Ε, έχω συναντήσει τον ε, Αμερικανό ομόλογό μου όταν έλαβε τα καθήκοντά του. Θεωρώ ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα εκτός από το ελεύθερο εμπόριο και στην πολιτική ατζέντα των Αμερικανών και για παράδειγμα και η μεταρρύθμιση των θεμάτων υγείας και θα υπάρξουν και πολλοί ανταγωνιστές. Δηλαδή πολλοί τομεί ανταγωνιστικοί με την εμπορική πολιτική. Μπορούμε όμως, όμως να συνεργαστούμε και εδώ οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ και η Προεδρία ώστε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα του εμπορίου. Μία επίσης ερώτηση έγινε, έγινε για τις σημαντικές μεταφορές τεχνολογίας και με τον τρόπο αυτό την μετρίαση των συνεπειών στην, ε, της του κλίματος. Είναι και αυτό σημαντικό να το δούμε παράλληλα με τον ιατρικό τομέα. Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησία και ιδίω δεν είναι όμως αποκλειστικά, είναι μια προϋπόθεση για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καθαρής τεχνολογίας και μαζί, όπως άλλες οικονομίες της αγοράς η, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι πρέπει να προστατεύονται τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και η μεταφορά τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες χώρες και εκεί η συμφωνία EPR έχει σημαντικό ρόλο αλλά πρέπει και να γίνεται και μια προσπάθεια διευκόλυνσης της μεταφοράς τεχνολογίας. Η Ένωση εξετάζει τρόπους διευκόλυνσης της μεταφοράς τεχνολογίας, ιδίως ε, clean tech. Το, για τον κύριο Φιέλνερ, ας μιλήσω σου ειδικά, αφού είναι συμπατριώτης μου. Συμφωνώ την ανησυχία σας σχετικά με τον προστατευτισμό. Πρέπει να είμαστε διαρκώς, να επαγρυπνούμε διαρκώς απέναντι σε τέτοιες τάσεις. Την δημιουργία δηλαδή νέων φραγμών στο εμπόριο. Δηλαδή να μην καταργούμε ορισμένους και δημιουργούμε άλλους τέτοιους φραγμούς όταν εισάγουμε νέα ε, ε, νομοθεσία. Να καθιστούμε ε, σαφές ότι δεν, δεν επιτρέπεται να γύρονται τέτοιοι φραγμοί και μέσα στις ε, χώρες μέλη. Όταν μίλησα για ε, τέτοια θέματα σχετικά με αγαθά υπηρεσίες και τεχνολογίες ε, προστασίας του κλίματος, αυτό εννοούσα. Τώρα για την Ινδονησία. Έχουμε συνεργαστεί σημαντικά με την Ινδονησία για να αναπτύξουμε μια ε, βιώσιμη διαχείριση των δασών. Δεν νομίζω όμως ότι η έγερση φραγμών στο εμπόριο είναι η λύση για την αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας. Σχετικά με την Νότια Κορέα και την αυτοκινητοβιομηχανία. Και εγώ βεβαίως είμαι φίλη του αυτοκινήτου. Όμως εξέφρασα πριν την προσωπική μου άποψη για την Σουηδία, για, την, ε, ναι, για τη χώρα μου. Πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με την ε, Νότια Κορέα σε ευρύτερο πλαίσιο. Να δούμε ότι έχουμε πλειονότητα τομέων όπου θα κερδίσουμε πολλά από μια τέτοια ε, Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Και ότι τα προβλήματά μας εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με την αυτοκινητοβιομηχανία θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Ακόμη και αν μείνουν απ' έξω από οποιαδήποτε νέα FTA. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα χρειαστεί να λύσουμε έτσι και αλλιώ. Χρειάζεται να κάνουμε δηλαδή την αναδιάρθρωση της αυτοκινητοβιομηχανίας μας. Δεν λέω ότι πρέπει να κλείσουμε όλα τα εργοστάσια διότι μπορούμε να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε την αυτοκινητοβιομηχανία μας και να εκμεταλλευτούμε και την ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε δηλαδή όλες τις νέες τεχνολογίες που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και άλλες τεχνολογικές λύσεις. Και αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό όταν μιλούμε για μια παγκόσμια Ευρώπη, ένα παγκόσμιο ρόλο της Ευρώπης και μια ανταγωνιστικότητα. Για την Κολομβία δεν είπατε, λέει κύριε Λούκας. Ναι, συγγνώμη, το ξέχασα. Ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας αποτελεί βεβαίω ακρογωνίο λίθο της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει ε, εντοπίω πολιτικό διάλογο για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτός ο διάλογο είναι αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας με την Κολομβία. Η πίεση και η βία που ασκείται κατά συνδικαλιστών στην Κολομβία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική ανησυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ένωση έκανε μια σχετική δήλωση στην διάσκεψη του Ιουνίου φέτος, η Ένωση παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και θεωρεί ότι ο διάλογος εξακολουθεί να είναι ο καλύτερος τρόπος για να ασκήσει επιρροή για την βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι μόνο στην Κολομβία αλλά και σε πολλές άλλες χώρες όπου σημειώνονται προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρώτα λοιπόν ε, διάλογος και όχι απομόνωση. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ εξ ονόματος όλων των μελών για τις ειλικρινείς και πλήρες απαντήσεις που δώσατε στα πλαίσια του χρήσιμου και ενημερωτικού διαλόγου. Για όλες και όλους εσάς που δεν υπήρχε χρόνος να δώσετε, να, να, να ε, κάνετε ερωτήσεις, ε, επισημαίνω ότι ο Υπουργός ήταν εδώ στις 3 η ώρα και χρειάστηκε να περιμένει στις 3 και 20 για να αρχίσει ε, η συνεδρίαση και να μπορείτε να συζητήσετε. Χρειάζεται να σας περιμένω. Ευχαριστώντας σας κύριε Υπουργέ, θα πω ότι και εμείς ως μέλη της Επιτροπής ε, θα έρθουμε στη Γενέβη ε, για την Υπουργική Διάσκεψη και ελπίζω ότι θα είστε σε επαφή και μαζί μας στη διάρκεια της διάσκεψης αυτής και θα μας ενημερώνετε για το τι γίνεται. Αυτό θα είναι σημαντικό πλεονέκτημα για μας, για να μπορούμε να παρακολουθούμε έστω και αν πρόκειται για ένα 20 λεπτό. Θα το εκτιμήσουμε ιδιαίτερο, ιδιαίτερα αυτό εάν το πράξετε. Σας ευχαριστώ και πάλι για την έλευσή σας εδώ και σας εύχομαι για την υπόλοιπη περίοδο μέχρι τέλους της Προεδρίας σας καλή επιτυχία. Υπουργός, σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να σας ξαναδώ σύντομα.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 κύριε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και με συγχωρείτε που σας καθυστερώ. Αν όντω πρόκειται να διακόψουμε τώρα τη συνεδρίαση, όμως θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια όσον αφορά τα πρακτικά της συνεδρίασης των συντονιστών. Μπορώ να τα κάνω τώρα. Δύο σημεία όπου μας εξέπληξε το γεγονός ότι αναφέρεται ότι υπάρχει συμφωνία. Σημείο 4.2 για τις ακροάσεις. Νομίζω ότι συμφωνήσαμε ότι τουλάχιστον δύο ακροάσεις θα μπορούσαν να συγχωνευθούν. του κυρίου Κάσπαρη για τις ε, κοινωνικές ε, και περιβαλλοντικές προκλήσεις του εμπορίου και για τις προκλήσεις της μεταφοράς τεχνολογίας. Στην απόφαση όμως, έτσι όπως αναφέρεται στα πρακτικά, βλέπουμε μόνο να αναφέρεται η πρόταση του κυρίου Κάσπαρη και όχι το θέμα της μεταφοράς τεχνολογίας όταν έχουμε να κάνουμε με κλίμα και εμπόριο στα πλαίσια της Κοπενχάγης. Ένα δεύτερο σχόλιο τώρα όσον αφορά τους εισηγητές. Σημείο 9 δεν νομίζω ότι αποφασίσαμε όντως, είπατε κι εσείς ότι συζητάτε το θέμα, όσον αφορά την ε, διανομή εκθέσεων για μηδέν βαθμούς στους προηγούμενους συζητητές τους, όσον αφορά τις ε, οικονομικές εταιρικέ σχέσεις, για παράδειγμα. Σημείο 9, επαναλαμβάνω. Ja, vielleicht zu dem letzten Punkt, Punkt 9. Wir haben Daniel Κάσπαρη, για το τελευταίο, για το 9. Χθε δεν λήφθηκε επίσημα απόφαση, γι' αυτό και μπορεί να τροποποιηθεί. Γιατί δεν λήφθηκε απόφαση, διότι τελευταία είχε γίνει μια συζήτηση σχετικά με το ότι για αυτέ τι ε, εκθέσει δεν επρόκειτο να δοθούν νέοι πόντι, νέοι βαθμοί. Και εγώ ενημερώθηκα. σαφώ αυτή ήταν η συμφωνία την προηγούμενη εβδομάδα. Και γι' αυτό συμφωνώ να το θέσουμε το θέμα αυτό την επόμενη φορά στην ημερήσια διάταξη των συντονιστών. Αλλά και την απόφαση που θα πρέπει να λάβουμε την επόμενη φορά με του συντονιστέ, ότι δηλαδή τα πράγματα όντω είναι έτσι όπω συζητήθηκαν και όπω έχουν σχεδιαστεί. Και νομίζω μάλιστα χθε έτσι το είδε και η πλειοψηφία. Δηλαδή, οι ε, εκθέσει οι οποίε προέρχονται από την προηγούμενη θητεία να παραμείνουν στα χέρια των ε, πολιτικών ομάδων που τι είχαν μέχρι τώρα ήδη έναντι 0 βαθμών. Συμφωνώ ωστόσο ότι θα πρέπει να συζητηθεί ξανά την επόμενη, στην επόμενη συνάντηση των συντονιστών. Και για την ακρόαση, δεν μιλούμε για ακρόαση που θα κρατήσει ολόκληρο το απόγευμα, αλλά για μήνυ ακρόαση. Και νομίζω ότι το θέμα αυτό αναφέρεται ακριβώ σε αυτό που λέτε. Δηλαδή στο ερώτημα πώ μπορούμε να συζητήσουμε για θέματα διευκόλυνση των εξαγωγών, ε, μεταφορά τη τεχνολογία ε, στην εξωτερική πολιτική, πολιτική περιβάλλοντο κλπ. κλίματο αλλά είμαι βέβαιο άλλωστε ότι περιλαμβάνεται στον τίτλο αυτό. Και νομίζω ότι στα πλαίσια αυτή τη μήνυα ακροάσεω ή και σε δύο μήνυα ακροάσει μπορούμε να ρίξουμε ιδιαίτερο βάρο στα θέματα αυτά. Να δούμε δηλαδή ποια μπορεί να είναι η συμβολή τη εξωτερική πολιτική σε διάφορου άλλου τομεί πολιτική. Και θεωρώ ότι το... στο θέμα αυτό όλε οι πολιτικέ ομάδε, αν εξετάσω τι ε, συζητήσει που έχουμε κάνει τα τελευταία πέντε χρόνια, έχουν να διδαχθούν πολλά πράγματα. Διότι υπήρξαν πολλοί συνάδελφοι που είπαν τα τελευταία πέντε χρόνια ότι η εμπορική πολιτική είναι καθαρή εμπορική πολιτική και δεν χρειάζεται να ανακατεύεται πουθενά αλλού. Όμω υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι φόρτωσαν στην εμπορική πολιτική πολλά άλλα πράγματα. Και είπαν για παράδειγμα ότι εάν έχει αποτύχει η αγροτική πολιτική θα πρέπει να διορθώσει τα πράγματα η εμπορική πολιτική. Αν έχει αποτύχει η περιβαλλοντική πολιτική πάλι να τα διορθώσει η εμπορική πολιτική και ούτω Ας δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς σε μία ή δύο μήνες ακροάσεις να εξετάσουμε το θέμα κάπως εγκύτερα. Και είναι το θέμα αυτό. Πραγματικά για τα επόμενα δύο-τρία χρόνια ποια μπορεί να είναι πραγματικά, ρεαλιστικά η συμβολή της εμπορικής πολιτικής σε άλλους τομείς πολιτικής. Εγώ είμαι ε, ευχαρίστως διατεθειμένος να υποστηρίξω δύο μήνυα ακροάσει για το θέμα αυτό. Yes, Σας καλύψαμε στα ερωτήματά σας. Βλέπω ξανά τα πρακτικά για τις ακροάσεις.